Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δύσκολο να το αποφύγει κανείς δεδομένου και του θέματος του περασμένου σημείου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα και άξιζε τον κόπο να γίνει αυτή η συζήτηση. Τώρα όμως χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση περνάμε στο σημείο 9. Αντιπροσωπεία του hoc των Επιτροπών Λίμπεντε Βεντρουά στο Παγκόσμιο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στη Γενέβη, η οποία διεξήχθη ε, στις 15 με 18 Δεκεμβρίου του 2019. Θα περάσουμε σε αυτό το σημείο της συζήτησης για να ακούσουμε ε, τι θα μας πούν τα μέλη ε, αυτής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο λόγω Φόρουμ. Ποια είναι η εμπειρία τους, η έκθεση τους και τα συμπεράσματα. Η κυρία Πιόρκ ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής, η οποία στενή εξ όσων γνωρίζω. Άρα θα την αντικαταστήσει κάποια άλλη συνάδελφο, σωστά τα λέω, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το είπατε προηγουμένω, λέει κυρία Ντουπον. Πρόκειται για την ad αντιπροσωπεία που είχαμε τρεις επιτροπές Λίμπε, Ντρουά και Ντέβε. Ε, πριν σα παρουσιάσω σύντομα την έκθεση, να ευχαριστήσω ρητά τη Γραμματεία και την ε, τη προσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωση στη Γενέβη για τη διοργάνωση, για την πλαισίωση και για τη συνοδεία ε, και την υποδοχή. Το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ήταν το πρώτο υπ' αυτή τη μορφή μετά ε, ε, την απόφαση ε, του κώδικα ε, για τους πρόσφυγες. Είναι πάνω από 25 εκατομμύρια οι πρόσφυγες παγκοσμίως και καλό ήταν που έγινε αυτή η συζήτηση για θέματα που τους αφορούν, στέγη, εργασία, προστασία γενικά. Η ε, αντιπροσωπεία μας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνεδρίαση όπου τα βασικά κράτη του Παγκοσμίου Φόρουμ για τους πρόσφυγες παρουσίασαν τις βέλτιστες πρακτικές τους, συμμετείχαν σε διάφορες συνεδριάσεις spotlight όπως τις λέγανε. Αφρική, Λατινική Αμερική ήταν τα κέντρα βάρους και είχαμε και θεματικές ενότητες, ας πούμε, η σχέση ανθρωπιστικής βοήθειας και ε, αναπτυξιακής πολιτικής. και ό,τι ξέχασα ή όσους ξέχασα θα τα συμπληρώσουν οι συνάδελφοι. Είχαμε πολύ, πολλές διμερές επαφές, κυρίως ε, ε, με το Συμβούλιο της Δανίας και της Νορβηγίας για τους πρόσφυγες, το Παγκόσμιο Δίκτυο. Την Τρίτη είχαμε ε, μια συζήτηση για την πράσινη υποδοχή των προσφύγων, για την μετακατάσταση και με την Oxfam, τη Διεθνή Επιτροπή Διδιάσωσης και πολλές άλλες εθνικές αντιπροσωπείες, Γερμανία, Καναδά, Ελβετία, Νίγηρα, ε, Ουγκάντα, Ρουάντα. Και επίσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ήπατη Αρμοστία. Το αποτέλεσμα γενικά του φόρουμ είναι πάνω από 800 ε, ε, υποσχέσεις κρατών, ΜΚΟ αλλά και ιδιωτών στα έξι θέματα που σας ανέφερα προηγουμένως για τη στήριξη των ε, προσφύγων και πρόληψη σειράξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως ασχολήθηκε με τη μετεγκατάσταση και τη συνέχιση των μέτρων που μέχρι τώρα εφαρμόζει ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια, για τις χώρες υποδοχής και για την αναπτυξιακή βοήθεια. Το επόμενο φόρουμ θα είναι το 2023. Στο τέλος ε, κάναμε και ένα δελτίο τύπου όπου ε, αναφέραμε τους στόχους μας και πάλι και τα αιτήματά μας και από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούμε να ε, εντείνουν τις προσπάθειές τους ε, να εντείνουν τις διεθνείς τους επαφές και να αναλάβουν τις διεθνείς υποχρεώσεις. Η αναπτυξιακή βοήθεια και η ανθρωπιστική θα πρέπει να συνεργάζονται, να προχωρήσουμε για το πακέλο ασύλου και μετανάστευσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρουμε στη σταθερότητα και στην ε, ε, ειρήνευση στις εμπόλεμες περιοχές για να χτυπήσουμε τη ρίζα του κακού της προσφυγιάς. Ευχαριστώ κύριε Τζιπόν. Η κυρία Μπιόρκ δεν είναι εδώ. Στα γερμανικά ο πρόεδρος. Ήταν πρόεδρος και εσείς ήσασταν επίσης μέλος. That delegation willing to make a point or contribution. Yes, I see. Λοιπόν, ε, θα είναι και άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν. Βλέπω ότι ζητείτε το λόγο. Η κυρία Σιλβάνα Γονσάλες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι γεγονός. Είχα την τιμή να είμαι κι εγώ μέλος της αντιπροσωπείας αυτής στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες. Συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Ντυπών για τα θέματα που εξετάσαμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν, και το διαπιστώσαμε και οι ίδιοι, ότι δεν τηρούνται ε, όλες αυτές οι υποσχέσεις κατάσταση, ή επανεκατάσταση ε, σε όλες ε, τις επαφές που είχαμε αυτό μας ζητούσαν να ε, ανταποκριθούμε στις υποσχέσεις μας. Ε, θέλω να πω και κάτι άλλο και το αναφέρει πολύ ωραία η έκθεση. Βέβαια να ευχαριστήσω ε, προηγουμένως ε, την γραμματεία της Επιτροπής μας αλλά και της Επιτροπής ΔΕΒΕ που ήταν μαζί μας και που ήταν πολύ ευαίσθητη στις προτάσεις που είχαμε εκπονήσει στην Επιτροπή ΔΕΒΕ. Τι θέλαμε, να εγγράψουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλη αυτή την κινητικότητα ε, και τη μετακίνηση πληθυσμών. Ε, λόγω κλιματικής αλλαγής υπάρχουν χώρες αναπτυσσόμενες που πλήττονται περισσότερο και έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Βλέπω ότι έχει ενταχθεί στην ε, έκθεση και θα πρέπει να προχωρήσουμε και να ε, ε, προχωρήσουμε στον ορισμό του κλιματικού πρόσφυγα. Ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει σε πολλούς και πολλές οργανώσεις δεν το κατανοούν, ούτε υπάρχει πουθενά στο διεθνές δίκαιο. Αλλά από την Ευρώπη εμείς πιστεύω έχουμε ευθύνη να ε, προωθήσουμε αυτό το θέμα και να δώσουμε προστασία στα εκατομμύρια των προσώπων που ήδη εντοπίζονται. Βέβαια, οι περισσότεροι είναι στο εσωτερικό της χώρας τους, αλλά πολλοί παίρνουν και τα σύνορα για κλιματικούς λόγους. Κάναμε διάφορες ε, συνεδριάσεις με οργανώσεις που ενέχονται πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα και ξέρω ότι διοργανώνεται μια τέτοια πλατφόρμα για τις θεομηνίες και τις επιπτώσεις τους. Υπάρχουν κάποιες χώρες τώρα που πρωτοστατούν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια αυτή και νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα, πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προσθέσουμε και αυτό στα συμπεράσματα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ οι δύο επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΝΤΕΒΕ για να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε προστασία στους ανθρώπους αυτούς που γίνονται πρόσφυγες λόγω ε, της κλιματικής αλλαγής και ε, υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια αυτή θα είναι εκατομμύρια. Ευχαριστώ κυρία Σιλβάνα μου στα γερμανικά τώρα, ο κύριος Μάρκαρτ, αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ε, τις σκέψεις σας και τις εμπειρίες σας. Βεβαίως, στα αγγλικά ο κύριος Μάρκαρτ. Ε, ήθελα να πω στην αρχή της συζήτησης. Um, ε, δεν έχει αλλάξει η... Ε, ε, δική μου εντύπωση. Θέλω να υπογραμμίσω τα όσα είπαν οι προλαλήσασες για τη σημασία ε, της συνεργασίας εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εκεί. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ΝΤΕΒΕ δηλαδή μαζί, εσωτερική και εξωτερική διάσταση. Φυσικά ε, για τη μετανάστευση και για άλλα θέματα για τους εκτοπισμένους. Και εξ ονόματος της Επιτροπής ΔΕΒΕ και του Κοινοβουλίου γενικότερα, τα σημαντικότερα για μας ποια είναι. Πρώτον, να συνεχίζουμε να προάγουμε και να προωθούμε πολυμερή συνεργασία για λύση βάσει κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου. Και έχουμε και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες τα ευρωπαϊκά κράτη, τα κράτη-μέλη της Ένωσης το έχουν υπογραμμίσει ε, το, και το έχουν υποστηρίξει. Θα πρέπει να εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τα θέματα αυτά και το θέμα της ε, ε, μετανάστευσης του εκτοπισμού για λόγους κλιματικής αλλαγής και χρειαζόμαστε καλύτερο καταμερισμό των ευθυνών όχι μόνο στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια, την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και ε, στο άσυλο και στην Ευρώπη και ε, γενικότερα. Θα πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτοι πρόσφυγες με την επανεγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια εκεί. Εχθές είδα ότι για κάποια κρατημέλη είναι πολύ εύκολο να έχουν μια ταχεία διαδικασία ενώ κάποια άλλα κράτη-μέλη έχουν υποσχεθεί και συγκεκριμένους χώρους για επανεγκαταστάσεις, αλλά οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ αργές. Ευχαριστώ κύριε Μάρκαρτ. Ο κύριος Καχέν, ήσασταν και εσείς μέλος της αντιπροσωπείας στη Γενέβη. Ναι, ναι. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ε, θα πρέπει και εγώ να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την ε, θαυμάσια και τέλεια διοργάνωση ε, ε, ήταν πολύ ε, καλές οι επαφές που είχαμε σε όλα τα επίπεδα. Είχαμε και εκπροσώπους των προσφύγων. Δεν άκουσα τις αρχικές τοποθετήσεις, δεν ξέρω αν το είπατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ήθελαν και εκείνοι να συμμετέχουν στις αποφάσεις που λαμβάνονται για εκείνους. Ε, και είναι καλό να έχουμε επαφές μαζί σου. μου έλειψαν εκεί οι χώρε, οι επίσημοι εκπρόσωποι. Ήταν λίγε οι χώρε, ήταν η Γερμανία και κάποιε άλλε και οργανώσει, αλλά όχι σε επίπεδο υπουργών. Και παρόλα αυτά μας λένε ότι στην Ευρώπη ιδιαίτερα είναι σημαντικό το πρόβλημα. Επίσης είχαμε ενδιαφέρουσες συνομιλίες με, ε, με τον Καναδά, την, ε, ε, τον Νίγηρα μάλλον, και για τη διαδικασία του Δουβλίνου το συζήτησαμε και χθε βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί το θέμα αυτό της επανεγκατάσταση. γιατί ο Νίγηρα που είχε συμφωνήσει για να φύγουν κάποιοι από τη Λιβύη και τα φρικτά βασανιστήρια. Η Γαλλία ε, είχε δεσμευτεί ότι μέσα σε δύο χρόνια θα πάρει 1.350 και πήρε μόνο 250 και άφησε τον Ήγερα στα κρύα του Λουτρού, ενώ η Γερμανία ανταποκρίθηκε στις υποσχέσεις της και όσους είχε πει ότι θα υποδεχθεί τους πήρε. Δεν ξέρω αν οι συμφωνίες αυτές είναι διμερείς ή πολυμερείς ή παγκόσμιες ε, γενικότερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θέμα της μετεγκατάστασης είναι πολύ ακαθόδες. Είδα και ένα πρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας και θα πρέπει να τονίσουμε ε, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των πόλεων για την κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική ε, ένταξη των μεταναστών. Είναι στην πρώτη γραμμή η Δήμη. Όταν φτάνουν οι μετανάστες, με νόμιμο ή μη τρόπο, δεν έχει σημασία, οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση. Οπότε θα πρέπει οι πόλεις να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στη διαδικασία λήψη απόφασης. Και η εκπρόσωπος, είπα, της αρμοστίας πραγματικά αποκρίθηκε θετικά. Το επόμενο φόρουμ θα γίνει το 2013 ακούσαμε προηγουμένως, αλλά το πρόβλημα είναι τωρινό. Και θα πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά για να ξεφύγουμε από αυτό που ονομάζουμε μεταναστευτικό πρόβλημα. Δεν είναι μεταναστευτικό το πρόβλημα, πρόβλημα υποδοχής είναι. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ανασκουμποθούμε και να κάνουμε πιο συχνές συναντήσεις, ίσως όχι σε επίπεδο γενική Γραμματείας του ΟΗΕ, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση και όχι μόνο εδώ στην Επιτροπή Λύπη, αλλά πάγια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Επίσης, άλλα ε, μέλη τη αντιπροσωπεία έχουν το λόγο. But I don't see them in the room. They are... Δεν τους βλέπω στην αίθουσα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να σχολιάσει. Αν όχι, συμπεράσματα, συμπεράσματα, όχι. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Έτσι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της μέρης σας διάταξης. Χαιρετίζουμε τα μέλη Ντέβε και Ντρουά που μοιράστηκαν ε, τις πληροφορίες αυτές μαζί μας. Yes. Mr. Chair, I'm sorry to... Με συγγνώμη που διακόπτω. Όπως ξέρετε, χτες το βράδυ στο Χανάο έγινε μία τρομοκρατική ενέργεια. Εννέα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Είχαμε μία συζήτηση για ε, τον εξτρεμιστή από που προέρχεται. Θα ήταν σκόπιμο ίσως να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή γιατί είναι μεγάλο το σοκ σήμερα στη Γερμανία. Έτσι αναγνωρίζουμε το τι συνέβη χτες το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και την υπόδειξή σας. Το είδα σήμερα το πρωί από τα μέσα που μας ενημερώνουν συνέχεια. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το σοκ. Χτες είχαμε μία συζήτηση και σε ένα από τα σημεία Τη συζήτηση είπαμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε τις εξελίξεις σε σχέση με την άκρα δεξιά που προβάλλει εγκλήματα μίσους. Εγκλήματα, όχι ρητορία μίσους. Και χτες ακούσαμε ορισμένα μέλη να εκφράζονται πολύ άσχημα. σε σχέση μια τρελή, με μια τρελή συμμαχία μεταξύ αριστεράς και Ισλάμ, σαν να πρόκειται για την πέμπτη φάλαγγα ε, μαζικής τρομοκρατίας, εγκλήματος και εγκλήματος στην Ευρώπη. Ωραία, ενός λεπτού σίγη παρακαλώ. Thank you all. Thank you. Σας ευχαριστώ όλους.